συμφωνία έγκαιρα. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ ολοκληρώνω. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο.